Δεν θα πω λοιπόν πάλι τα ίδια. Θα ήθελα να υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων περισσότερο. Θα ήθελα να καθορίσω το πλαίσιο στο οποίο θα κάνουμε τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Πρόκειται για τρία στοιχεία τα οποία παίζουν ένα ρόλο για αυτό το νέο μέσο. Το πρώτο είναι ένα θέμα στρατηγικής. Πρόκειται για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά της Ένωσης. Πρέπει να είναι συνεπής η πολιτική, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις άλλες πολιτικές mainstreaming, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο και πώς θα το συνδυάσουμε με αυτό το νέο μέσο EIDHR. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για πολλές μη ΚΑΠΑΟΜΙΚΡΟΝ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και στα άλλα μέσα, αλλά και στον πολιτικό διάλογο με τις ε, διάφορες χώρες, να μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι εναλλακτική στον πολιτικό διάλογο, αλλά είναι συστατικό του πολιτικού διάλογου. Δεύτερον, στο νομοθετικό τομέα είναι ένας κανονισμός εδώ, πώς θα πρέπει να εγκριθεί για να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ε, κατάλληλο όργανο για να μπορεί να προωθεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχέση με τι άλλε χώρε. Επίση πρέπει να δούμε πώ θα ενταχθεί στον δημοσιονομικό ε, στο δημοσιονομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες της Ένωσης. Και κάτι τρίτο συγκεκριμένο, πρακτικό. Πώς θα εφαρμόσει επιτόπους διάφορες χώρες η, πολιτική, η Ένωση την πολιτική της, πώς θα την ε, αντιληφθούν οι χώρες όπου εφαρμόζεται. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες πολιτική και στις τοπικές συνθήκες, που είναι περίπλοκες. Διότι οι διαδικασίες μας είναι βαριές, είναι περίπλοκες. Και γι' αυτό ορισμένες μη καπαόμικρον δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα μέσα της Ένωσης. Άρα ίσω να μην μπορούν να αξιοποιήσουν και αυτό. Βεβαίω, όλα αυτά τα προβλήματα δεν θα τα επιλύσουμε μέσω τη έγκριση αυτού του κανονισμού αλλά πιστεύω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να συμπεριληφθεί στη δέσμη μέτρων μα. Καλωσορίζω λοιπόν του τρει προσκεκλημένους μα που προέρχονται από, διαφορετικά, από διαφορετικούς οργανισμούς. Όλοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Ο Ζωάν Πολ είναι εδώ και πολύ καιρό ανταποκριτής της εφημερίδας Λουσουάρ και είναι σύμβουλος της Επιτροπής για την προστασία των δημοσιογράφων και του Παρατηρητήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ο δεύτερος εκπρόσωπος και κυρίως ο τρίτος εκπρόσωπος που με ενδιαφέρει που είναι από την Τινησία. Χαίρομαι πολύ που είναι δυνατόν να δώσουμε τώρα αμέσω ε, με τη σειρά που θα καθορίσει ο Πρόεδρος αν με ακούσει, αν με ακούσει ο Πρόεδρος να πει πώς θα δώσει το λόγο στους τρεις εμπειρογνώμονες. Με ποια σειρά. Ο κύριος Μαρτός, λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις περισσότερο πολιτικής φύσεως και όχι τόσο τεχνικής. Πιστεύω πως διανύουμε μια φάση που σηματοδοτείται από μια υποχώρηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτή η πρωτοβουλία σημαίνει ότι θα πρέπει να αρθούμε στο επίπεδο αυτής της πρόκλησης που είναι πολύ σοβαρή καθώς και μια ε, σταθερή πολιτική βούληση στο βαθμό όπου όλα τα προγράμματα για τη δημοκρατία και την ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αμφισβητηθούν. Να θυμίσω την πρόσφατη ε, φυλάκιση κάποιων ανθρώπων στην Αίγυπτο που ήταν εκεί για να εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα και μάλιστα γερμανικής εθνικότητας. Ε, σημαίνει δηλαδή την ανάληψη ρίσκου, κινδύνου ε, για τα προγράμματα αυτά. Και επίση ανταγωνισμό όλο ένα και μεγαλύτερο όσον αφορά την αποφασιστικότητα των πολιτικών προτύπων σε ολόκληρο τον κόσμο, α πούμε στα αραβικέ και μουσουλμανικέ χώρε όπω το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία δαπάνησαν πάνω γύρω στο 1 δι δολάρια σε προγράμματα στήριξη των Ισλαμιστικών κινημάτων. Και η Κίνα αναπτύσσει ένα κοινό μάλλον ε, σχολές δημοσιογραφικές που σίγουρα δεν είναι αυτές που εμείς θα ε, σκεφτόμασταν όταν, ε, όταν μιλάμε για ελεύθερη έκφραση και δημοσιογραφία. Να πούμε τώρα ότι η εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη της δημοκρατίας στο παρελθόν ήταν πολύ σημαντική. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και του 90 η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε πολύ αποτελεσματικά με τα βάση στην Χιλή και στην Νότια Αφρική και εγώ παρακολούθησα από πολύ κοντά αυτές τις δύο ε, προσπάθειες που θεωρούνται ως πραγματικές επιτυχίες της δημόσιας διπλωματίας αλλά και της στήριξης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε να αποκομίσουμε χρήσιμα διδάγματα Καταρχήν, βαθιά γνώση της πολιτική κατάστασης των λόγω χωρών. Πράγμα που δεν ίσχυε όταν ε, πρόκειται για άλλε χώρε που παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια των ετών. Επίσης, ε, σε ξεκάθαρε επιλογές για στήριξη δημοκρατικών ε, κομμάτων αποκλειστικά, αποκλείοντα του υπόλοιπου. Δηλαδή, δεν προσπαθούσαμε να έχουμε σχέσει με του κυβερνητικού θεσμού απαραίτητο, πράγμα το οποίο διευκρίνησε ξεκάθαρα πιανού την πλευρά παίρναμε και υπέρ τίνο πράγματος. Εξαιρετικά επιλεκτική στήριξη δηλαδή. Για παράδειγμα, όταν, όσον αφορούσε τη στήριξη του τύπου, δεν ε, στηρίζαμε γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εκείνα τα οποία παίζανε ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο στη μετάβαση. Ας πούμε, του Weekly Mail Guardian, που στην ε, στην Νότια Αφρική ή αντίστοιχα τη Χιλή που στήριζαν την μετάβαση και όχι δεν υποστηρίζαμε γενικά τα μέσα μαζική ενημέρωση και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Επίσης επρόκειτο για στρατηγική στήριξη όπου λαμβάνομαι υπόψη την ε, ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω χωρών και για παράδειγμα στις δύο χώρες αυτές στηρίξαμε θεσμούς, ερευνητικά κέντρα ακαδημαϊκά κέντρα τα οποία ήταν, στην ουσία λειτουργούσαν ως ε, υποκατάστατα των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση ακαδημαϊκών ε, συστημάτων. Επίσης αυτό που ήταν σημαντικό σε αυτές τις χώρες ήταν η ανάγκη να διατηρήσουμε αυτονομία και ανεξαρτησία απέναντι στα κράτη, τα κράτη-μέλη και τις, και τις δικές τους λογικές και συμφέροντα. Και πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνοχή όσον αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της σε σχέση με αυτές τις χώρες. Η συνοχή αυτή θα έπρεπε, έπρεπε επίσης να έρχεται από τα από πάνω, δηλαδή να έχουμε το πιο ψηλό κοινό παρονομαστή και όχι το πιο χαμηλό, το μικρότερο. Η συνοχή είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική και η συγκρότηση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι σε κάποιες ε, αραβικές χώρες δεν μπορεί να σταθεί πλέον. Δεν μπορούμε όπως παλιά να ασκούμε πολιτικές όπου ταυτόχρονα ε, ε, παίζαμε με τις αυταρχικές κυβερνήσεις ενώ υποστηρίζαμε και τα δημοκρατικά κινήματα. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει την γραμμή της και τη στήριξή της σε αυτούς τους φορείς της δημοκρατικής γνήσης, της δημοκρατικής μετάβασης και όχι απλά μια συμφιλίωση ανάμεσα τώρα στα αυταρχικά συστήματα και τους δημοκράτες. Επίσης θα πρέπει να δουλέψουμε κατά τη γνώμη μου πάνω σε ένα σύστημα που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ταχύτητα στις παρεμβάσεις. Πολύ συχνά υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ανάμεσα στις τα γεγονότα επιτόπου και τη δυνατότητα ανταπόκρισης των μέσων. Σημαντικό είναι να μπορούμε να δούμε τα κριτήρια κατανομής, οι διαδικασίε να είναι πιο ευέλικτε και πιο εύκολε, υπό δημοκρατικό έλεγχο πάντα φυσικά, αλλά πιο απλέ, ώστε να είναι μέσα στον κύκλο των γεγονότων. Εφόσον θέλουμε δηλαδή να συνεργαστούμε με τοπικές οργανώσεις, ώστε ακριβώ να μην φαίνεται σαν να είμαστε μια, ε, μια εξουσία που θέλει να παίξει, να επηρεάσει υπερβολικά τη χώρα, πράγμα το οποίο θα σήμαινε ότι κάποιοι δικαιούχοι ευρωπαϊκής βοήθειας ε, θα, σήμαινε, θα, θα, ε, θα χαρακτηρίζονταν ως υποστηρικτές του συστήματος έτσι ώστε οι μεταβάσεις να γίνονται ε, χωρίς να είμαστε πολύ κοντά στους κύκλους εξουσίας στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. είναι ο Κάρλος Φερνάντες που είναι εκτελεστικός διευθυντής ε, για την εταιρική σχέση για τη δημοκρατία από το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα σχολιάσει την πρόταση της Επιτροπής ως έχει και τις τροπολογίες. Παρακαλώ, για πέντε λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα είμαι σύντομος. Γενικά μιλώντας, από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών, ο κανονισμός που συζητάμε τώρα και οι τροπολογίες φαίνεται να είναι στο σωστό δρόμο. Και αυτό συμβαίνει γιατί η εντύπωση που έχουμε σχηματίσει είναι ότι το μέσο με το οποίο ασχολούμαστε στο νέο κανονισμό είναι πιο συνεκτικό όσον αφορά τους στόχους και με ποιο τρόπο θα συνδυάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επίσης, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος για να υπογραμμιστεί ο ρόλος των ίδιων στις αλλαγές. είναι κάτι που όσο και να το υπογραμμίσουμε δεν φτάνει. Επίσης, επειδή υπάρχει τάση να ενισχύουμε, να σταθεροποιούμε κατά κάποιο τρόπο τις δυνατότητες που έχει το μέσο να δρά σε πιο δύσκολες χώρες και να υποστηρίζει τους αγωνιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εδραιώνονται τέτοιοι μηχανισμοί στήριξής τους και επίσης έτσι ενισχύεται και η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν να μπορεί να δράσει σε έκτακτες περιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι βοηθάει την πολιτική συζήτηση. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και σίγουρα ενισχύθηκαν όλα αυτά με την Αραβική Άνοιξη. Υπάρχουν όμως και κάποια θέματα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα όσον αφορά τη, τον κανονισμό του EDHR. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη συμπληρωματικότητα. Δεύτερον, την ελαστικότητα. Και τρίτον, δημοκρατικός έλεγχος και διαχείριση του μέσου. Όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα, το είπαν και άλλοι πριν από μένα, συζητιέται παντού. Ως πολιτική αρχή είναι ζωτική σημασία, όπως και συνοχή, και δεν θα πρέπει να παραμεριστεί. Το ζήτημα που παραμένει είναι το κατά πόσο ο κανονισμός είναι και ο κατάλληλος τρόπος για να συζητήσουμε την ε, συμπληρωματικότητα και πώς θα εφαρμοστεί αυτή. Σε κάθε χώρα είναι διαφορετικά, άλλο, είναι προγραμματικά προγράμματα. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κανονισμός. Γι' αυτό θέλουμε να ενθαρρύνουμε τόσο την Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο να μην ε, κάνουν μνήα σε πολλά σημεία σε κανονισμό, αλλά να γίνει μια γενική σύσταση προκειμένου να υπάρξει μια γενική εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι μέσα υπάρχουν για τη συμπληρωματικότητα. Βλέπετε μερικές φορές προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα τα οποία μοιάζουν ή συγκρίνουμε διάφορα μέσα, αλλά συνήθως είναι πιο σημαντικό να δούμε ποια είναι η συμπληρωματικότητα με το DCI, για παράδειγμα, με κάτι άλλο. Επίσης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερικές φορές δείχνει να μην είναι συνεπής, αλλά αυτό έχει να κάνει με την πολιτική που βρίσκεται από πίσω. Πρέπει να υπογραμμίσουμε πάντως τη δυνατότητα που έχει το μέσο αυτό να αντιμετωπίσει έκτακτες περιπτώσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι οι προτάσεις οι οποίες βρίσκονται στο τραπέζι είναι καλές. Πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανθρώπινα δικαιώματα, μεσοδιευκόλυνση, απλοποίηση των διαδικασιών για κάτω από 100.000 ευρώ. Όλα αυτά είναι θετικά. Πρέπει να παραμείνουν όμως τα όρια για την απευθείας κονδύλια όσον αφορά τις έκτακτες καταστάσεις. Η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να δράσει στις χώρες αυτές, περιορίζοντας την χρηματοδότηση σε προτάσεις που είναι κάτω των 100.000 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μπορεί να κάνει κάτι σε έκτακτες περιπτώσεις. Το κύριο βέβαια ζήτημα είναι η διαδικασία. Πώς θα διασφαλιστεί ο έλεγχος και η ευελιξία. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τα ποσά, έχει να κάνει με τη διαδικασία. Το τελευταίο ήταν ο δημοκρατικός έλεγχος, που βέβαια συνδέεται με το προηγούμενο. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα του σώματος αυτού, για παράδειγμα, να ελέγχει την διαχείριση του EDHR. Πρέπει να δούμε και με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό. Εμείς δεν είμαστε σίγουροι για το ότι η συζήτηση γύρω από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις είναι ό,τι καλύτερο. Το σώμα εδώ πρέπει να μπορεί να ελέγχει και γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται παραπάνω σκέψη πάνω σε αυτό. Αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ντίλια Ρέμπαε, ιδρυτικό μέλος της, ε, την, της ε, Ένωσης για τη Δημοκρατία και της ε, ε, ε, ε, δημοκρατικές εκλογές της Τινησίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε την καλή διάθεση να ακούσετε την κοινωνία πολιτών της Τινησίας που είναι ο κύριος ενδιαφερόμενος της συζητήσης. Εμείς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούμε από αυτό το μέσο. Είμαστε η κύρια δύναμη επιτόπου που συνεχίζει να μάχεται για μια ουσιαστική δημοκρατία στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα να σας παρουσιάσω την ένωσή μας η οποία δημιουργήθηκε πριν από λιγότερο από ένα χρόνο μετά την Επανάσταση το Μάρτιο. Έχουμε 2.600 μέλη. Έχουμε γραφεία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, στις Τινησίες, 25 γραφεία και επίσης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένε Πολιτείε, το Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι για να παρατηρούμε εκλογές. Έχουμε παρατηρήσει εκλογές στις 23 Οκτωβρίου. Μετά τις εκλογές αυτές οργανώσαμε συναντήσεις εκλογέων εκλεγμένων για θέματα που θα συζητήσει η Συντακτική Εθνοσυνέλευση και την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε την πρότασή μας για τη δημιουργία μιας νέας δομής που στόχο θα έχει να διεξαγάγει τις προσεχείς εκλογές. ή χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι περί αυτού πρόκειται στη συζήτηση αυτή. Τι ωφέλη θα μπορούσαν να χορηγήσουν αυτές ε, οι χρηματοδοτήσεις στις ε, χώρες σε φάση εκδημοκρατισμού, ελπίζω, ταχαίως εκδημοκρατισμού. Βεβαίως έχουμε και τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες αξίες. Και βεβαίως θέλουμε η Τινησία να μπορέσει να γίνει πλήρως λειτουργική δημοκρατία. Ξέρουμε ότι στη χώρα μας τα συμφέροντα της Ευρώπης ε, είναι επίσης σημαντικό να έχει καλούς γείτονες. Άρα είναι σημαντικό να υπάρξει δημοκρατία στην Τινησία και για την Ευρώπη. Δεύτερον, η εικόνα που έχουν οι πολίτες μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια εικόνα ουδετερότητας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας εκεί να υπάρχει αυτή η εικόνα αντικειμενικότητας και ουδετερότητας γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε ποιοι σας χρηματοδοτούν και ορισμένες φορές έχουμε αρνηθεί χρηματοδοτήσεις λόγω του χορηγού. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας επιτρέπει κάπως να αποκαταστήσουμε την ισορροπία διότι πάρα πολλά χρήματα δίδονται αυτή τη στιγμή στην Τινησία, πολλές χρηματοδοτήσεις, πολλές δυνάμεις προσπαθούν να παρέμβουν. Είναι λοιπόν ένα αντιστάθμισμα σημαντικό η χρηματοδότηση της Ένωσης προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών. Ποια είναι τα μειονεκτήματα, τα αρνητικά που διαπιστώνουμε για αυτούς που λαμβάνουν αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα, δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια πού πρέπει να απευθυνθούμε, πού πρέπει να κάνουμε αίτηση. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Τα μέσα βεβαίως υφίστανται, αλλά δεν είναι πάντα προσαρμοσμένα για τις ανάγκες αυτών των ε, προσφάτων ε, ενώσεων που δημιουργήθηκαν μετά την Ένωση. Για παράδειγμα, πρέπει να πληρούν διάφορα κριτήρια που πολλές φορές ε, δεν είναι δυνατόν. Επίσης, οι διαδικασία σας δεν είναι αρκετά ταχείε. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει αναγκαία ευελιξία και ετοιμότητα σε σχέση με άλλους χρηματοδότες κυρίως. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν, τόνισα, περισσότερη ευελιξία περισσότερη ετοιμότητα και δυνατότητα αν κάποια γραμμή του προπολογισμού δεν μπορεί να μας χρηματοδοτήσει να μπορούμε να περάσουμε σε άλλη. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να ήμουν σαφής και θα απαντήσω φυσικά στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η Σκιώδης τώρα. Η να ίσως η πρώτη. Όχι. Δεν θέλετε το λόγο. Είσαστε οι πρώτοι σκιώδεις που βλέπω τουλάχιστον. Η κυρία Γκόμες χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για την παρουσίασή τους εδώ και για το ότι είναι στη διάθεσή μας να απαντήσουν τις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ και τον Αλεξάνδερ, ο οποίος ανέλαβε και την πρωτοβουλία να σας προσκαλέσει εδώ. Είναι πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή. Θέλω να σας ρωτήσω όμως κάποια πράγματα ακόμα. Για τον κύριο Μάρτος. Στα καθήκοντά σας, στο Human Rights Watch, έχετε διαπιστώσει να κινητοποιείτε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις οργανώσεις δηλαδή που περιλαμβάνονται σε εσά έχετε διαπιστώσει ότι πάνε χώρες, πάνε στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, εκεί δηλαδή όπου με τη διάσκεψη των Παρισίων η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε να καταρτήσει τα μέσα ενημέρωση. Έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα μέσα ενημέρωσης που προωθούν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πλουραλισμό, την ε, ανοχή. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα επίπεδο γενικής στήριξης, ρυθμιστική, δεντολογική, που και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και που κάποιος πρέπει να αναλάβει. Οπότε σας ρωτάω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει και αυτή να συνεισφέρει. Όμως θέλω να ξέρω, εσείς και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας, Έχετε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει τον ρόλο της. Ε, έχει δραστηριοποιηθεί δηλαδή για να χρησιμοποιήσει τη δικιά σας εμπειρία και να καταρτιστούν έτσι και συνάδελφοί σας στις ε, διάφορες χώρες. Κύριε Νάντες, μπορείτε να μας πείτε γιατί η κατεξουσιοδότηση πράξης δεν είναι καλό μέσο για να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Τέλος κύριε Ριμπάη. σημείωσα τόσα είπατε ότι δεν υπάρχει ελαστικότητα, ταχύτητα. Ρωτάω λοιπόν, έχετε την αίσθηση ότι στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τινησία υπάρχει ένα focus point, ένα γραφείο τέλο πάντων το οποίο να μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, το οποίο να μπορείτε να υποβάλλετε σχέδια, προγράμματα στα πλαίσια της δράσης σας. Και πώς αξιολογείτε εσείς τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάτε για την ουδετερότητα απέναντι στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία ή απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε εννοείται ή όταν το NDMA έχει παίξει το ρόλο του για να καταρτήσει παρατηρητές στην Τινησία. Εσείς πώς βλέπετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε όργανα όπως για παράδειγμα το NDI και τόσα έχει κάνει. Με συγχωρείτε, ξέχασα να πω. Δύο λεπτά παρακαλώ, είναι ο χρόνο ομιλία, ξέχασα να το πω. Δύο λεπτά η κυρία Φρανσίσκα Τσάμπτον. Ωραία, θα ήταν καλύτερα να είχαμε μιλήσει προηγουμένω. Επιτρέψτε μου μία ερώτηση. Είπατε ότι είναι κυρίως θέμα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά μήπως νομίζετε πως είναι θέμα πολιτικής βούλησης ε, ή είναι θέμα κανονισμών είναι θέμα προσωπικού γιατί είναι πάντα μια ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε. Είναι θέμα δηλαδή εφαρμογής ή θα έπρεπε κάτι να αλλάξει ο κανονισμός ή κάποιο άλλο κείμενο για να γίνουν ευκολότερα τα πράγματα. Το δεύτερο και αν υπάρχει επαρκές προσωπικές, ε, προσωπικό επιτόπου ποιος είναι υπεύθυνο, ποιος μπορεί να είναι ο συνομιλητής των δικών μας των υπηρεσιών. Αν αυξήσετε δηλαδή το προσωπικό σας, θα μπορούσατε να λύσετε τα προβλήματα αυτά πρόσβασης πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις. Μία πρόταση ο Κόμις Λάμστορφ. Να έχει ρήμα η πρότασή μου, λέει ο κύριος Λάμστορφ. Να έχει, λέει ο κύριος Μπρόκ. Μια ερώτηση στο μέσο αυτό έχουμε και την παρατήρηση των εκλογών, δηλαδή τη μέρα της ψηφοφορίας. Η οργάνωσή σας βεβαίως ασχολείται και εκείνη με το θέμα αυτό. Θα θέλαμε όμως να μπορούμε να παρακολουθούμε τον πλήρη εκλογικό κύκλο, δηλαδή όλη την προεκλογική περίοδο να παρατηρούμε, να στηρίζουμε τη δημοκρατία. Ερώτημα λοιπόν προς τους τρεις και επανέρχεται σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρτός, η Ένωση θα έπρεπε να είναι πιο επιλεκτική δηλαδή να βοηθάει τις δυνάμεις που είναι υπέρ της μετάβασης ή να είναι αυστηρά ουδέτερη. Μιλήσατε για επιλεκτικότητα. Δηλαδή θα πρέπει να στηρίζουμε κάποιους και άλλους να μην τους στηρίζουμε. Αυτό δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα με την εικόνα αντικειμενικότητας και ουδετερότητας που θα πρέπει να έχουμε. Δεν είναι κίνδυνος αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Παρακαλώ τους εμπειρογνώμονε να είναι πολύ σύντομοι γιατί χρειαζόμαστε και άλλα 10 λεπτά για να συζητήσουμε πολύ σύντομα το θέμα της Συρίας. Παρακαλώ. Πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι προγράμματα χρηματοδοτεί στις αραβικές χώρες η Ένωση για να είναι πλήρης απάντησή μου. Ξέρω ότι πρόσφατα, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ενδιαφέρουσα διαβούλευση για τη Ρωσία που έδειξε πώς πρέπει να δουλεύουμε. Το προσωπικό του γραφείου της Ένωσης ε, στη Μόσχα συνεργάστηκαν μαζί μας και με τους ε, Ρώσους ε, δημοσιογράφους ούτω ώστε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Και με δική μας πρωτοβουλία στηρίξαμε και άτομα που ήταν θύματα επιθέσεων που σχετίζονται με κάποια κέντρα εξουσίας. Ήταν πολύ αποτελεσματικό το πρόγραμμα αυτό, ιδιαίτερα για κάποιο Μοσχοβίτη δημοσιογράφων. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντέδρασε γρήγορα. Και κατά την συνάντηση κορυφής απευθυνθήκαμε και στην Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων για να μάθει τι ε, αιτήματα είχαμε υποβάλει στον ε, Ρώσο εισαγγελέα για περιπτώσεις ε, δολοφονίας δημοσιογράφων. Τέτοιου τύπου ενέργειες πρέπει να κάνουμε σε συνεργασία με τις τοπικές αλλά και διεθνείς Επιλεκτικότητα. Εγώ, επειδή θέλω να έχω συγκεκριμένα αποτελέσματα, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ποιον να στηρίξει η Ένωση και ποιον όχι. Ποιες πολιτικές ή κοινωνικές δυνάμεις, κυρίως σε χώρες σε περίοδο μετάβασης. Αλλά δεν χρειάζεται να περιζόμαστε σε αυτό, όπως είπε η κυρία Γκόμες. Μπορούμε να βοηθήσουμε την ενίσχυση των θεσμών. Για παράδειγμα, τους νόμους για τα μέσα, την ε, μετατροπή των κρατικών ΜΜΕ σε ελεύθερα ΜΜΕ, να συνεργαστούμε δηλαδή και με τοπικές αρχές και με θεσμούς, ακόμη και κυβερνητικούς. Πολιτικά όμως θεμελιώδες είναι να καταδείξουμε ποιο είναι το μήνυμα της Ένωσης. Στηρίζουμε δηλαδή την μετάβαση στην οποία τον κύριο ρόλο παίζουν οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ευχαριστώ. Ο επόμενος. να <clears throat> συνεχίσω μετά από την ε, απάντηση αυτή. Δουλεύουμε για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προωθήσουμε την ουδετερότητα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα ουδετερότητα γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε υπέρ κάποιων αρχών δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό ιδιαίτερα μέσω του μέσου που μα επιτρέπει ακριβώ να το πετύχουμε αυτό. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση τη Άννα Γκόμε για τι κατεξουσιοδότηση πράξη. Είναι βέβαια τεχνική η συζήτηση, άρα και βαρετή. Πάντω, έχουμε κάποια ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον ορισμό τη κατεξουσιοδότηση πράξη. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ουσιώδη ζητήματα. Όμω, η συζήτηση μέχρι τώρα όσον αφορά το μέσο γίνεται να χρησιμοποιούνται κατά εξοδότηση πράξεις για τις ετήσιες ε, πράξεις. Με αυτά είναι ουσιώδη πράγματα, έχουν να κάνουν με την πολιτική μας. Δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε εσείς, αλλά συγχρόνως είναι περίεργο πώς να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή να είναι και για μη ουσιώδη, αλλά από την άλλη να είναι για αυτά τα θέματα που μας φαίνονται ουσιώδη. Τώρα, η κατεξουσιοδότηση πράξη δεν θα έδινε περισσότερο έλεγχο στο κοινοβούλιο και δεν θα το επέτρεπε να έχει περισσότερη δύναμη. Για δύο λόγους. Γιατί, Γιατί το κοινοβούλιο, βέβαια είναι συζητήσιμο αυτό, το βάζει μέσα σε όλη την ε, διαδικασία, αλλά μένεται σε περιορισμένες επιλογές. Ή κυρία ή τίποτα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δει αυτό κανείς. Πάντως, για μένα, αλλά και οι συνάδελφοί μου το ίδιο πιστεύουν, το κύριο θέμα θα ήταν ότι μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων δεν μπαίνει μόνο το Κοινοβούλιο στην όλη εικόνα, αλλά και το Συμβούλιο. Και εδώ είναι που έχουμε επιφυλάξεις. Είναι αυτό που προσπαθούσα να πω και πριν, ότι πολλά από τα θέματα που συζητάμε εδώ μπορεί να εξεταστούν με έλλειψη συνοχής. Εγώ πιστεύω ότι η κατεξουσιοδότηση πράξης μπορούν να το φιλτράρουν αυτό, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο θετικό. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι να έχει ισχυρό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχει και να ακούει το EDHR να λογοδοτεί για το τι κάνει. Αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι ο καλύτερος τρόπος είναι αυτές οι κατεξουδότηση πράξεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εσείς. Δεν ξέρω ποια είναι δικιά σας γνώμη, αν είναι αντίθετη. Θέλω να απαντήσω κι εγώ για τις δύο μεγάλες ερωτήσεις που μου θέσατε. Πρώτα απ' όλα για την ουδετερότητα της Ευρώπης. Η ουδετερότητα έχει να κάνει και με άλλους οργανισμούς, το NGI και τα λοιπά. Στην Τινησία πάντως, τόπου... είναι γεγονός. Η αμερικανική χρηματοδότηση ε, δεν ε, γίνεται αντιληπτή θετικά τουλάχιστον από ένα μεγάλο μέρος. Για το MEP, για παράδειγμα, όπου είχα εγώ συμβόλαιο, αναγκάστηκα να πω όχι. Γιατί δεν θα πέρναγε. Άρα υπάρχει αυτός ο περιορισμός που τον έχουμε και εμείς υπόψη μας και έχουμε να κάνουμε με αυτόν αναγκαστικά. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν ε, Παρεβαίνει στις επιλογές μας, εντάξει. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε πράγματα τα οποία δεν δέχεται βάση. Όσον αφορά τώρα την ευελιξία των κονδυλίων που χορηγούνται. Εκτός μικροφώνου κάνει μια ερώτηση ο πρόεδρος. Τι εννοώ όταν λέω η βάση. Ενώ οι παρατηρητές Πάντα, κάθε φορά και πολλές φορές συνέβη αυτό μετά τις εκλογές λιγότερα, κάθε φορά που έδινα συνέντευξη, η πρώτη ερώτηση που μου κάνανε, α, πώς χρηματοδοτήστε, πάντα, πώς χρηματοδοτήστε. Και αν έλεγα Ενωμένες Πολιτές της Αμερικής, τελείωσε, θα είχαμε χάσει την αξιοπιστία μας. Απλώς και μόνο γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, την πολιτική τους, την χρησιμοποιούν αλλού, όχι τόσο για την, την Ισία, πάντως η την Ισία πλήττεται από αυτό. Μιλάω λοιπόν τώρα για την ευελιξία των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο που άλλοι είναι πιο δραστήριοι. Πέρσι πριν 10 μήνες περίπου, όπου και πάλι μου κάνετε τη τιμή να μ' ακούσατε, είχα ζητήσει επιγόντως πόρους για να καταρτιστούν οι παρατηρητές. Δυστυχώς, τα κονδύλια αυτά δεν έχουν πληρωθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν άπειρα τέτοια παραδείγματα που δείχνουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση επιτόπου ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δραστηριότητα. Αν, ας πούμε, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέντε μέρες, από τότε μέχρι τότε θα είναι η κατάρτιση αυτή. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε τις διαδικασίες ε, ψηφοφορίες που δεν, είναι στα δικά μας τα χέρια. Και γιατί να κάνουμε αυτή την κατάρτιση με διαδικασίες που δεν υπάρχουν ακόμα. Θα ήταν προτιμότερο να το κάνουμε για δύο-τρεις μέρες. Δεν έγινε όμως, οπότε δεν έγινε καν η κατάρτιση καθόλου. Για μικρές διαδικασίες λοιπόν ισχύει αυτό. Έπειτα το σημερινό σύστημα αξιολόγηση. Έχετε τρία χρόνια εμπειρία για οργανώσεις οι οποίες φτιάχτηκαν μετά την Αραβική Άνοιξη. Πού να τη βρουν τα τρία χρόνια εμπειρίας μετά ή για άλλα προγράμματα που έχουμε επιτόπου. Εμείς ένα χρόνο έχουμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά που ζητάτε δεν είναι εφαρμόσιμα στις δικές μας τις οργανώσεις. Θα μπορούσα να σας μιλάω για ώρες για αυτά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Για να σας πω ότι αυτές οι διαδικασίες δεν προσαρμόζονται, ενώ χρήματα υπάρχουν και στην Τινησία υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να είναι οι χώρες του κόλπου, δεν μπορώ να έχω αποδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλες οργανώσεις Εμεί θελήσαμε να είμαστε πολιτικά ουδέτεροι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε τι δικέ μας πολιτικές απόψεις, αλλά αυτές δεν τι διαφημίζουμε. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν οργανώσεις οι οποίε είναι πολιτικοποιημένες δικαιωμά και αυτές αμέσως έχουν τα χρήματα που τους χρειάζονται όταν τα χρειάζονται. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο για μας γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την ευελιξία. Άρα δεν έχουμε αυτή την αλλακτική λύση. Ελπίζω να απάντησα. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Αλλά προηγουμένω να σας πω ότι αυτά τα παραδείγματα που μας δώσατε είναι πολύ χρήσιμα. Δείχνουν γιατί πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι να μπορούμε να επηρεάσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλιώς οι, επιβάλλονται οι γραφειοκρατικές δομές. Και όταν διαπιστώνουμε ότι σε τέτοια πράγματα ζητάμε τρία χρόνια εμπειρία, δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι αστείο στην ουσία αυτό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Μία φράση κύριε Λάμπστροφ, διότι οι διερμηνείς έχουν ήδη ξεπεράσει το ωράριό τους. Ε, ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για την παρουσία σας που μας μιλήσατε. Πιστεύω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ. Πρέπει να δούμε οπωσδήποτε το θέμα αυτό των κατεξιοδότηση πράξεων, αλλά το τελευταίο παράδειγμα ήταν πολύ συγκεκριμένο. Καταδεικνύει ότι το μέσο αυτό πρέπει να γίνει ακόμη πιο ευέλικτο, αλλά βεβαίω πρέπει οπωσδήποτε να περάσει και στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρω, ξέρω. Γι' αυτό Πρέπει να υπάρξει αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία για να μπορεί να δρά συντομότερα. Πρέπει να δούμε συνολικά το όλο πακέτο, την όλη δέσμη μέτρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ε, χρήσιμη. Ευχαριστώ κύριε, Πρόεδρε, κύριε Λάμσδορφ που ε, ευχαριστήσατε και εκ μέρους του Προέδρου. Και σίγουρα σε ψηλό και κόμις. Και έχουμε λίγα λεπτά. Έχουμε εδώ τον κύριο Έλκα Ουζουτάλο που είναι επιματάρχης για τη Μέση Ανατολή. Παρακαλώ σύντομα να μας πείτε τι συνέβη. Και να μας πείτε πώς έχει ε, αντιδράσει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ. Γιατί πρέπει να έρθετε εδώ μπροστά. Παρακαλώ, αρχίστε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάθαμε για το νέο αποτρόπαιο επεισόδιο, το φόνο αμάχων στην Αλγερία. Αυτό αποδεικνύει ότι η κατάσταση είναι μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της βίας που στοχεύει επί τούτο τους αμάχους. Η κατάσταση αυτή είναι στο προσκήνιο όλων των ε, προσπάθειων που μπορεί να κάνει και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η κυρία Άστον, ούτω ώστε μαζί με τους ε, εταίρους μας παγκοσμίως να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Όμως υπάρχει μια αντίφαση όλες οι κύριες δυνάμεις φαίνεται να λένε ότι συμμορφούνται προς το σχέδιο ΑΝΑΝ αλλά εξακολουθούν να συμβαίνουν στην πράξη διαφορετικά πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπου δεν προχωράει το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις και δολοφονία μάχων στη Χάμα, ενώ μιλάμε, θα υπάρξει μια δήλωση της κυρία Άστον, όπου πέρα από την καταδίκη αυτού του φρικαλαίου εγκλήματος και των φόνων καλεί για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση όχι μόνο αυτού του εγκλήματος αλλά και των προηγουμένων που συνέβησαν στη Χούλα πριν από μόλις δύο εβδομάδες. Καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα να δράσει ενωμένα για να καταστεί δυνατό να υπάρξει μια πολιτική διαδικασία. Μόλις χθε το βράδυ συναντήθηκε στη Κωνσταντινούπολη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Αντιτρομοκρατικού Φόρουμ σε μια συζήτηση για τη Συρία. Συζήτησε και με Ρώσους εκπροσώπους ε, αρχές της εβδομάδας διότι η Ρωσία παίζει ρόλο κλειδί για να απεμπλακεί η κατάσταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ξέρετε ότι σήμερα ο Κόφι Ανάν ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και υπάρχουν κάποιες προσδοκίες ότι θα υποβληθούν από τον ε, ίδιο κάποιες νέες προτάσεις για να προχωρήσει το θέμα για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή του σχεδίου ανάν. Όπως αναφέρεται στον τύπο μπορεί να συμπεριλάβει προτάσεις για να δημιουργηθεί ένα είδος ε, ομάδος πυρήνα εθνών για να υπάρξει απεμπλοκή της κατάστασης. Το θέμα αυτό βεβαίω προσετέθη στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε η κυρία Άστον θα είναι παρούσα για να σε ενημερώσει για τις επαφές με τους διάφορους εταίρους και να σε ενημερώσει για τις διάφορες συναντήσεις στι οποίε έχει πάρει μέρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαστε όλοι ιδιαίτερα θλιμμένοι. Δεν έχει υπάρξει βέβαια εξωτερική επιβεβαίωση για τη Χάμα αλλά για τη Χούλα είδαμε τις φωτογραφίες 30 άτομα τα οποία εκτελέστηκαν ψυχρό. Είναι τρομερά αυτά τα γεγονότα, είναι σαν αυτά που συνέβησαν στα Δυτικά Βαλκάνια πριν από 10 χρόνια. Θα ήθελα να καταλάβουμε ότι το κλειδί είναι ε, η Ρωσία. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών έκανε κάποια σχόλια της Ρωσίας και μου το ανέφερε ένας πρέσβης της ε, του Αραβικού Συνδέσμου ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα να υπάρξει μια Συρία χωρίς τον Ασάντο Πρόεδρο. Υπάρχει μια αλλαγή στη στάση της Ρωσίας. Αν είναι δυνατόν να υπάρξει η Ρωσία χωρίς τον Άσαντο Πρόεδρο, θα κινηθεί η Συρία ή συγγνώμη, η Ρωσία ώστε να αναιρέσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η στάση των κρατών μελών. Τι νομίζει η κυρία Άστον ότι μπορούμε να κάνουμε για να πιέσουμε ακόμη περισσότερο τη Συρία να αντιληφθεί την Ρωσία, να αντιληφθεί λοιπόν η Ρωσία ότι πρέπει να καταλήψει τη Συρία, τη σύμμαχό τη, να καταλήψει το καθεστώ ε, του Μπαθ. Να απομονωθεί η Συρία, να απομονωθεί και από το Ιράν. Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι έχει πολύ ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα στη χώρα του κόλπου και τη συνεργασία με, το, με τις χώρες του Συμφώνου Συνεργασίας του Κόλπου και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ένα καθεστώς του οποίου οι πράκτορες ε, με ασυδοσία δολοφονούν γυναίκες και παιδιά. Είναι περίπλοκη βεβαίως η κατάσταση, η αντίσταση βεβαίως επίσης δεν είναι άγια, αλλά όλες οι ενδείξεις φαίνεται να καταδεικνύουν ότι έχει επιτρέψει στις, στις πολιτοφυλακές της των αλαβητών να πηγαίνουν από χωριό σε χωριό, να τρομοκρατούν και να δολοφονούν γυναίκες και παιδιά. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας κατά τη γνώμη μου. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα πολιτικά. Ξέρουμε που είναι το κλειδί για μια αλλαγή. Υπόθηκε, είναι στη Ρωσία, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για αυτούς. Σίγουρα δεν θα στείλουμε ανεπάνδρωτα αεροσκάφη drones να γκρεμίσουν τα σπίτια των ηθινόντων του καθεστώτος. Υπάρχουν όμως κάποιοι τομείς όπου δεν έχουμε ακόμη διακόψει τις οικονομικές επαφές. Υπάρχουν πτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Συρία είναι κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες και οι συριακές ε, αερογραμμές. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα ως επόμενο βήμα να διακόψουμε όλες τις πτήσεις από και προς τη Δαμασκό από κράτη μέλη της Ένωσης. Από τη γνώμη μου θα ήταν κάτι συγκεκριμένο και θα μπορούσαμε να κλείσουμε και τα λιμάνια μας προς όλα τα συριακά σκάφη για να ε, σταματήσει κάθε επαφή με τη Συρία. Η κυρία Γκόμες. χωρίς να δημιουργηθεί πολιτικό πρόβλημα, να πω ότι συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος Στάνοκ. Το κλειδί είναι η Ρωσία. Και πιστεύω πως η Κίνα θα ακολουθήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τον τρόπο να είναι πιο αποτελεσματική, να πιέσει και να κατονομάσει τη Ρωσία. Thank you. Frau Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ε, και έχουμε αυτό το αίσθημα της ανημπόριας. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να κάνουμε κάτι έναντι της Ρωσίας, να αλλάξει δηλαδή ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα συμφέροντά τους οι Ρώσοι. Ξέρουμε τι θα θέλανε, για παράδειγμα οι Ρώσοι, να διευκολύνουμε τις βίζες. Θα είμαστε εντεθειμένοι να κάνουμε λοιπόν κάποια αντίμετρα έναντι του κυρίου Πούτιν να του πούμε κύριε Πούτιν θα διευκολύνουμε τη διαδικασία για τις προξενικές θεωρήσεις εάν σταματήσεις να υποστηρίζεις τον Άσαντ. Είναι σημαντικό νομίζω. Δεν αρκεί το να λέμε ποιος φταίει για να ντραπεί. Πρέπει κάτι να κάνουμε για να πιέσουμε τη Ρωσία. Και το δεύτερο, για την αντιπολίτευση, έχουμε επαφές με το SNC, αλλά δεν κατάφερε το τελευταίο εξάμεινο ή ένα άμυνο να ενοποιηθεί η ενα Να συμμετέχουν δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια και επιτόπου μαχόμενοι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ισχυρό ρόλο ούτω ώστε να μην χρησιμοποιεί και να χειραγωγεί κάποια τμήματα της αντιπολίτευσης, κάποια δύναμη. Πρέπει να δράσουμε επιτόπου, να υπάρξει ενοποίηση της αντιπολίτευσης αυτό μας ζητούν. Και τη δυνατότητα επίσης να συνενώνονται και εκτός Συρίας οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς εκπροσωπεί το SNC. Δεν λέω ότι δεν έχει πια καμία αντιπροσωπευτικότητα, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, ομάδες. Πρέπει να απευθυνθούμε και σε αυτές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολουθούμε μια κατάσταση απαράδεκτη. Τα νέα που μας έρχονται μιλάνε για 68 νεκρούς, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι μαχαιρώθηκαν από αυτή την πολιτοφυλακή του Πρόεδρο ΣΑΤ. Τα έχουμε πει και ξαναπεί Ακούσαμε τι είπανε και οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, ε, χτες στην Κωνσταντινούπολη. Η στάση των Ρώσων είναι απαράδεκτη. Διότι θέλουν να συμπεριλάβουν το Ιράν, για παράδειγμα. Πάντω η δήλωση την επόμενη εβδομάδα που θα κάνει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να αναλάβει μια πιο συγκεκριμένη δράση ώστε ο πρόεδρος της Συρίας να καταλάβει ότι αυτά τα οποία έγιναν στην Αίγυπτο, στη Λιβύη μπορεί να το συμβούν και του ίδιου. Είναι απαράδεκτο να συνεχίζουμε με σταυρωμένα τα χέρια να βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση αδυναμίας απέναντι σε δολοφονίες σαν και αυτές που λαμβάνουν χώρα στη Συρία. Νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πρόεδρε, πρέπει να είναι σε θέση να βάλει τη φαντασία του να δουλέψει και να βρει τρόπους να δράσει για να βοηθήσει την κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι η διάσκεψη αυτή που έγινε πρόσφατα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία δεν ήταν αποτελεσματική, έτσι όπως τα θέλαμε τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Σα Yes. Ε, um, Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο γιατί θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε απαντήσεις σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα και φυσικά θα διαβιβάσω όλες αυτές τις ερωτήσεις στην ύπατη εκπρόσωπο όταν θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ε, αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια το θέμα της αλλαγής της ρωσικής θέσης δυστυχώς δεν είδαμε καμία αλλαγή ε, νωρίτερα ήδη μίλησαν και έδωσαν την εντύπωση ότι για αυτούς η Συρία θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς τον Ασάντ. Δεν ήταν όμως ξεκάθαρη και ιδιαίτερα με τις ε, ενέργειές τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν υπήρξε αλλαγή. Από την οικονομική πλευρά θα ήθελα να πω και να θυμίσω ότι έχουμε 15 φορές ε, παρατείνει το καθεστώς των κυρώσεων που ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο και πάνω στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ίσως να ληφθούν περαιτέρω σχετικά μέτρα ε, γι' αυτό εργαζόμαστε. Επίσης πριν δύο μέρες συμμετείχαμε σε μια διεθνή συνάντηση στην Washington περί ε, για να προσπαθήσουμε να έχουμε και άλλους εκτός της Ένωσης ε, που θα ακολουθήσουν το καθεστώς των κυρώσεων γιατί είναι σημαντικό να έχουμε συμμάχους που προβαίνουν στη λήψη παρόμοιων μέτρων ώστε τα μέτρα αυτά να είναι αποτελεσματικά. Εν γέννη, για να πείσουμε την ε, Ρωσία, έγινε μια ε, διάσκεψη κορυφή. Ε, είπατε, είπατε εκπρόσωποι ήταν στη διαρκή επαφή μαζί του για να προσπαθήσει να το προωθήσει το θέμα και έγιναν και, και μάλλον συνεχίζονται αυτές οι συζητήσει. Σε σχέση με την αντιπολίτευση, δυστυχώς είναι κατακαιρματισμένη, δεν έχει μπορέσει να καταλήξει σε μια ισχυρή ενωπημένη βάση να σας πω όμως το εξής, μιλάμε με όλους, όλες τις, διαφορετικές, τις διάφορες ομάδες όχι μόνο αυτήν του EAS. Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε μήπως μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε αυτές τις ομάδες, γιατί έγινε αυτή η αποτυχημένη προσπάθεια από τον Αραβικό Σύνδεσμο στις 6 Απριλίου. Ε, προσπαθούμε λοιπόν μήπως τα καταφέρουμε και έχουμε και μόνιμη επαφή με τον Αραβικό Σύνδεσμο γι' αυτό. Οι προσπάθειε λοιπόν συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα και την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε και περισσότερα από την ίδια την ύπατη εκπρόσωπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερω επειδή ήρθατε τόσο σύντομα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το προσωπικό μου αίσθημα είναι ότι ότι πρέπει να τονίσουμε ότι το σχέδιο Ανάν δεν έχει πλέον καμία αξία. Είδαμε ότι όχι μόνο τους εκτελούν, αλλά μετά τους ποδοπατούν κιόλας. Είδαμε τις εικόνες. Δεν υπάρχει πια καμία συμφωνία δεν μπορούμε πλέον να τη χρησιμοποιούμε ως πρόσχημα. Ευχαριστώ πολύ.